έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη θετική στάση της. Ευεπιστώ ότι αυτό το χαρτοφυλάκιο θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε λοιπόν με αυτή την πορεία μας.